και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να ε, προχωρούμε με τα παραδοτέα επί των θεμάτων που θίξατε και εσείς σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, τους ε, επιτρόπους. Στο πέρας της ε, συζητήσεως έχουμε έξι ψηφίσματα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση. Θα λάβει χώρα η ψηφοφορία αύριο στις 12.30. Βάσει τη ημερήσια διάταξη, λοιπόν, οδηγούμεθα ή στι προφορικέ ερωτήσει προ την Επιτροπή σχετικά με την κρίση στην Καμπανία στον τομέα των αποβλήτων. Θα δώσουμε πρώτο το λόγο στου συγγραφεί ε, πρώτα απ' όλα την ε, κυρία Όουκεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, ε, Επίτροπε Ποτότσνικ. Φαίνεται ότι η Κομισιόν καμιά φορά είναι συνεπέστατη στη δράση της. Καλό είναι η δράση αυτή να είναι και ορατή. Ελπίζω ότι απόψε θα πάρουμε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί αν δεν γίνει και τώρα τίποτα, δηλαδή αν δεν επιβληθούν αυστηρές ποινές στην Ιταλία, όλο και θα προσκρούμε στο πρόβλημα αυτό, γιατί υπάρχουν τεράστια προβλήματα ε, αποβλήτων. Και όταν κάποιος αποκομίσει την εντύπωση ότι κανείς δεν νοιάζεται για την αποκομιδή των σκουπιδιών, τότε οι καταστροφές θα είναι μεγάλες. Για την Ιταλία τώρα. Ξέρω ότι εδώ δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενη η Ιταλική κυβέρνηση, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αρχίσει να αντιμετωπίζει. Τι ωραία χώρα και να θαυτεί από τα σκουπίδια. Τα βουνά των σκουπιδιών αυξάνονται και η κατάσταση διαρκώς χειροτερεύει. Ο πληθυσμός στην Ιταλία δεν πρέπει να επιβαρύνεται άλλο με το πρόβλημα αυτό. Αντίθετα, θα πρέπει να αναπτύξει ένα καλό πρόγραμμα αποκομιδής. και πολλοί δραστήριοι πολίτες θα συμμετέχουν ως μέρος της λύσης χωρίς να ε, ποινικοποιούνται. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των σκουπιδιών αν δεν συμμετέχουν και οι πολίτες. Θα τους εντάξουμε και υπάρχουν πολλοί που είναι πρόθυμοι να ενταχθούν. Και ο στρατός και η αστυνομία μπορούν να χρησιμεύσουν. Δεν χρειάζονται μόνο για να καταπιέζουν τον πληθυσμό και να, να δημιουργούν προβλήματα στις τοπικές κοινότητες, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τους πραγματικούς εγκληματίες, τα μεγάλα, ε, τις μεγάλες βιομηχανίες, τις μεγάλες μονάδες στην Ιταλία που θέλουν να απαλλαχθούν φθηνά από τα σκουπίδια, η μεγάλη γκάγκστερ, η μαφία. Ε, πρέπει λοιπόν στην Ιταλία να πιάσουν ε, σοβαρά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για δύο λεπτά, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού πήγε το φθινόπωρο στην Ιταλία και εκεί ε, συναντήσαμε τον πρόεδρο της ε, Καμπανίας ε, της περιφέρειας αυτής και το ρωτήσαμε γιατί δεν είχε επιληθεί ακόμα το πρόβλημα αυτό και μας απάντησε μας λέγοντας ότι πρόκειται για ένα πολιτικό πρόβλημα. Αυτό λέει πολλά γιατί θα μπορούσε να είχε πει άλλα πράγματα που μπορούσαν πει ότι είναι ένα τεχνικό πρόβλημα, πρόβλημα λογιστικής φύσεως ή οικονομικό πρόβλημα. Όχι, είπε πως το πρόβλημα είναι πολιτικό. Το πρόβλημα είναι ότι απουσιάζει η πολιτική βούληση και αυτή η έλλειψη της πολιτικής βούλησης έχει οδηγεί έχει σαν αποτέλεσμα η Ιταλία να μην αναλαμβάνει τις δεσμεύσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με την οδηγία αποκομιδής των απορριμμάτων. Είναι λοιπόν η απουσία πολιτικής βούλησης που έχει σαν αποτέλεσμα τον Οκτώβριο να μην έχουν εφαρμοστεί οι βελτιώσεις που απέτυσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον, οποίο η Ευρωπαϊκή, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα λάβει στα χέρια της κάπο σχέδιο ε, διαλογής και διαχωρισμού των απορριμμάτων στην Ιταλία. Οι αρχές ε, θέλουν να συγκαλύψουν όλα αυτά κρατώντας τα μυστικά. Αλλά εμείς στη δική μας ε, αντιπροσωπεία, στη δική μας ομάδα απαιτούμε ε, να ζητήσουμε να υποστηριχθούν οι Ιταλοί οι οποίοι θέλουν να πράξουν σωστά. Ε, θέλουμε οι υπόλογοι να διηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αλλά για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να αρνηθούμε οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι να πρέπει να πληρώσουν. Τέσσερα λεπτά η κυρία Μέρκιες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Με την Επιτροπή Αναφορών πήγαμε πέρσι στην Καμπανία, στην Άπολη, για να δούμε η διεισόμαση την κατάσταση επιτόπου. Να δούμε πώς ακριβώς είχαν τα πράγματα όσον αφορά αυτήν την επίγουσα κατάσταση ε, των ε, αποβλήτων ε, θέμα το οποίο αποτελούσε κεντρικό σημαντικό μέλημα πολλών αναφερομένων και πολλών αναφορών που έφτασαν στην Επιτροπή Αναφορών. Ε, είδαμε ε, καταστάσεις ε, πολύ διαφορετικές. Είδαμε, ας πούμε, τόπο αποκομιδής και εναπόθεσης σκουπιδιών στα, στους πρόποδες του Βεζουβίου, σε μια προστατευόμενη φυσική περιοχή. Ε, επίσης είδαμε περιπτώσεις ε, όπου ε, καίγονται τα σκουπίδια σε κέντρα καύσης μας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι υπήρχαν πολιτικά προβλήματα και επομένως ζητήσαμε να συναντηθούμε με εκπροσώπους των πολιτών και των πολιτικών έτσι ώστε να ακούσουμε διαφορετικές απόψεις αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε ακόμα να μιλήσουμε με όλο τον κόσμο έτσι ώστε ε, να καταλάβουμε εάν τελικά υφίσταται ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο ε, διαχείρισης ε, σύμφωνα με τους ε, πολίτες με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή μας ε, λένε ότι έχουν χτυπήσει όλες τις πόρτες της επαρχίας, της περιφέρειας, της πόλης, ε, του Δήμου, ε, της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά χωρίς καμία απάντηση. Γι' αυτό λοιπόν στράφηκαν σε εμά. Εμείς θελήσαμε να τους ακούσουμε, γιατί θέλαμε να καταλάβουμε τι περιμένουν από εμά, πώς θέλουν να συμβάλλουμε στην επίλυση της κρίσης στην περιοχή τους. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μην ε, ε, να μην σκοτώσουμε την ελπίδα αυτών των ανθρώπων, την ελπίδα που έχουν να αποθέσει στα χέρια μας. Ε, βεβαίως δεν μπορούμε εμείς να ανασηκώσουμε τα μανίκια μας, να ανασκουμποθούμε και να πάμε να καθαρίσουμε αυτές τις περιοχές οι οποίες πνίγονται κάτω από τόνους σκουπιδιών, αλλά πρέπει να, να μάθουμε ποιο είναι το προβλεπόμενο σχέδιο, ποιες είναι οι προβλεπόμενες προθεσμίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να στραφεί προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προτίθεται να επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα ε, στην ε, ε, χώρα αυτή. Με ποιο τρόπο θα παρέμβει ή προτίθεται να παρέμβει η Επιτροπή. Ξέρω ότι πρόκειται για δική σας αρμοδιότητα κύριε Επίτροπε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιες έρευνες σε σχέση με το πώς, ποιες θα είναι οι περιοχές στις οποίες θα γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών, εάν θα είναι προστατευόμενες και περιοχές κτλ. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα των ε, ε, μαφιόζικων οργανώσεων που ασχολούνται με τα σκουπίδια. Ε, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ή να βρεθούν τρόποι να γίνουν σεβαστές οι οδηγίες μας. Επίσης, με ποιο τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τα ίδια τα κράτη-μέλη. Τα σκουπίδια δεν είναι πρόβλημα μόνο, θα πρέπει να τα δούμε και σαν ευκαιρία. Η καμπανία θα μπορούσε να γίνει παράδειγμα ε, ε, ανακύκλωσης. Θα πρέπει να βρούμε το θάρρος να αποκλείσουμε και να ε, ε, θέσουμε εντελώς εκτός νόμου τις ανεξέλεγκτες χώματερες. Ευχαριστώ πολύ για δυόμιση λεπτά η κυρία Μπιτζότο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση που η καμπάνια και η η πόλη της Νάπολης αντιμετωπίζει είναι γνωστή πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε να ασχοληθεί επανειλημμένα με το ζήτημα αυτό απέναντι σε αυτήν την παράδοξη κατάσταση ε, που είναι τριτοκοσμική πλέον ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ε, ποιες ε, είναι οι ευθύνες της Ιταλίας σε σχέση με, τον, με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ποια είναι τα οικονομικά ή άλλου είδους πρόστιμα τα οποία ε, θα μπορούσε η Επιτροπή να ε, επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην καμπανία θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των σκουπιδιών Ξέρετε κύριε Επίτροπε, όταν αναφερόμαστε σε επικίνδυνες επίγουσες ε, καταστάσεις, ε, ε, αναφερόμαστε σε καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να περιμένουν. Όταν όμως μια τέτοια επίγουσα κατάσταση επιμικίνεται επί μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε κάτι δεν λειτουργεί καλά. Θα πρέπει <clears throat> να υπάρξει ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο διαχείρισης, συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων βεβαίως ένοχοι για την ε, λόγω ακριβώς της πλήρους αδυναμίας τους ε, να ενεργήσουν σωστά ε, είναι η τοπική πολιτική κοινωνία. Ξέρουμε ότι στον κύκλο των σκουπιδιών πολλοί είναι οι ένοχοι ε, στην πόλη, στο Δήμο, στην επαρχία, ε, σε ε, όλα τα επίπεδα. Αλλά βεβαίως δεν μπορεί να φταίει η κεντρική κυβέρνηση. Η κεντρική κυβέρνηση η οποία έχει στείλει, αναγκάστηκε να στείλει το στρατό και προημερών αλλά και σε άλλη χρονική στιγμή. Ε, αναγκάστηκε να το κάνει γιατί ε, τα προβλήματα υγείας και τα προβλήματα σχετικά με την βία που προκαλούσε η όλη κατάσταση ήταν πάρα πολύ ε, σημαντικά. όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ευθύνη για την κακή διαχείριση ε, της ε, κατάστασης, ε, ευθύνη λέγω, έχουν η πόλη και η επαρχία της Καμπανίας, καθώς επίσης και η διασυνδέσεις που παραδοσιακά έχει με τις εγκληματικές οργανώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος Ποτότσνικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έπεσαν την προσοχή μου και την προσοχή των υπηρεσιών μου σε αυτό το σημαντικό θέμα. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε έναν ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της κατάστασης των αποβλήτων στην Καμπανία, όπως έδειξε η έκθεση που ενέκρινε η Επιτροπή ε, το περασμένο Απρίλιο. Το Κοινοβούλιο παίζει πραγματικά ένα σημαντικό ρόλο εδώ και έχει αναλάβει πλήρως αυτό το ρόλο. Αμέσως μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το Μάρτιο του 2010 η Επιτροπή ρώτησε τις ταλικές Αρχές τι είδου μέτρα είχαν λάβει ή προγραμματίσει ούτως ώστε να συμμορφωθούν με αυτή την απόφαση του δικαστηρίου. Μετά από αυτό η Επιτροπή είχε διάφορες επαφές και συναντήσεις με τις ταλικές Αρχές και πιο πρόσφατα ε, ε, κατά την ε, στις 22 Νοεμβρίου του 2010 και την επίσκεψη της ε, αντιπροσωπείας της ε, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι οι Ιταλικές αρχές ακόμα έχουν ε, πολύ δρόμο μπροστά τους ώστε να εκτελέσουν την απόφαση του δικαστηρίου. Ιδιαιτέρως θα πρέπει πρώτον να παρατείνουν τις δυνατότητες διαχείρισης αποβλήτων και να ενισχύσουν σε όλη την ε, καμπανία και θα πρέπει να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης για τα αστικά απόβλητα λαμβάνοντας υπόψη τους μεταξύ άλλων την, ε, τις προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων. Η Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη με τα μέτρα που έχουν ε, ανακοινώσει οι τελικές αρχές μετά την ε, απόφαση του δικαστηρίου, γιατί ακριβώς δεν περιλαμβάνουν ένα λεπτομεριακό χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τις εργασίες για την ε, δημιουργία των υποδομών. Πιστεύουμε ότι το σχέδιο διαχείριση των αποβλήτων για την καμπανία θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρω με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θα πρέπει να δίδει προτεραιότητα στη μείωση των αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους και επίσης να εξασφαλίζει την εφαρμογή ξεχωριστής συλλογής των αποβλήτων στο σύνολο της περιφέρειας και να παράσχει στην καμπάνια τις απαραίτητες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης για την διάθεση και αποκομιθή των απορριμμάτων σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα και αυτό για πάνω από 7 εκατομμύρια στερεών αποβλήτων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει μία ανάλυση πριν, ληφθούν, πριν ληφθεί η απόφαση για το ποιος είναι ο πιο ασφαλής τρόπος διάθεσης των αποβλήτων. Εάν δεν υπάρξει ένα αποτελεσματικό πλάνο διαχείρισης, η Επιτροπή θα επανέλθει στο δικαστήριο και θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων. Γι' αυτό θα πρέπει να αξιολογήσουμε το πρόγραμμα διαχείρισης που οι αρχές της καμπανίας έχουν υποβάλει προλίγου ε, πρόσφατα στην Επιτροπή και θα πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά την έγκριση και την εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Η απόφαση για το κατά πόσο θα πρέπει να αρχίσουν οι διαδικασίες επιβαραβάση κατά της Ιταλίας θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο του σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων και το χρονδιάμαρμα εφαρμογής των μέτρων που έχουν σαν σκοπό να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή με ένα πιστικό τρόπο. Ε, σε σχέση με τις υπάρχουσες χωματερές, η Επιτροπή ε, ξεκίνησε μια σχετική έρευνα και ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να αναφέρουν για την λειτουργία των χωματερών του Τερτσιάνο και Τιλτσιάνο. Ε, εκκρεμεί ακόμα η απάντηση των Ιταλικών αρχών και αυτή τη στιγμή στη Λάβη η Επιτροπή θα την αξιολογήσει. Στη φάση αυτή η Επιτροπή δεν έχει προφανή στοιχεία για μια παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περιβάλλοντος. Το γεγονό ότι η χωματερή βρίσκεται σε ένα χώρο προστατευόμενο ε, δεν συνιστά αυτό καθ' αυτό μια παραβίαση της κοινωτικής νομοθεσίας ε, εφόσον βεβαίως εφαρμόζονται άλλες διατάξεις του νόμου και οι αρμόδιες αρχές ε, διενεργούν μια σωστή αξιολόγηση του περιβάλλοντος και εφαρμόζουν τα αναγκαία αντισταθμιστικά μέτρα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μέτρων του σχεδίου διαχείρισης Αποπλήτων στην Καμπανία, το 88 ε, εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για τέτοιου είδου προγράμματα. Ε, το, 49% ε, συγχρηματοδοτήθηκαν από την ERDF. και βεβαίως ένας επιβαρυντικός παράγων Ε, είναι η, ήταν ε, ε, οι, οι, συνθήκες. Εν μια 140 εκατομμύρια ευρώ και 50% από αυτά πάλι συγχρηματοδοτήθηκαν από το ERDF και δόθηκαν σε σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων. Ωστόσο μετά την κρίση, από τη, μετά την κρίση που ξέσπασε η Επιτροπή αποφάσισε να λάβει επιπρόσθετα μέτρα τους ώστε να εξασφαλίσει την σωστή αξιοποίηση των πόρων. Τον Ιανουάριο του 2005 ε, θεωρήθηκαν ε, μη εκλέξιμα τα μέτρα αυτά για την συγχρηματοδότηση. Ε, και η Επιτροπή ενημέρωσε το 2007 τις Ιταλικές Αρχές ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή περαιτέρω συγχρηματοδότηση. Το λειτουργικό πρόγραμμα 2007-2013 στην Καμπανία προβλέπει μια συνολική επένδυση 270 εκατομμυρίων ευρώ και πάλι το 50% συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο ε, Ανάπτυξης. Ε, οι επενδύσεις αυτές υπόκεινται ε, στην προϋπόθεση ότι οι Ιταλικές αρχές θα εγκρίνουν ένα ε, σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή. Αύριο θα δημοσιευθεί η έκθεση για την εφαρμογή της θεματικής στρατηγικής για την ανακύκλωση των αποβλήτων. Αυτή η έκθεση δείχνει σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών μελών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των αποβλήτων και δείχνει ξεκάθαρα ότι με μια σωστή στρατηγική διαχείριση των αποβλήτων οι χωματερές μπορούν να μειωθούν και να φτάσουν σε μηδενικό επίπεδο και με μεθόδους κομποστοποίησης και ανακύκλωση μπορεί σημαντικά να βελτιωθεί η κατάσταση. Ε, και με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται επίση θέσει εργασία και αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα, ενώ μειώνονται οι αρνητικέ περιβαλλοντικέ επιπτώσει ε, από τα απορρίμματα. Ελπίζω λοιπόν ότι η κρίση αυτή θα μετασχηματιστεί σε μια αληθινή ευκαιρία για τι αρμόδιε αρχέ μέσω τη εκπόνηση ε, ενό σχεδίου ε, διαλογή και συστήματος ανακύκλωσης των αποβλήτων στην Καμπανία. Η Επιτροπή ελπίζει το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων στην Καμπανία να είναι αξιόπιστο και να υπάρξει ένα σύστημα αποτελεσματικής υποδοχή, υποδομής και εγγυήσεις ότι το σχέδιο αυτό θα εφαρμοστεί. Εάν δεν γίνει αυτό, η χρηματοδότηση θα διακοπεί. Ε, βρίσκομαι στη διάθεσή σας για Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους αγορητές εξονόμητος των πολιτικών ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με την ε, κυρία Ματσόνη από το ΕΛΚ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε τον Επίτροπο γιατί ε, θύμισε ότι η Επιτροπή Αναφορών έδωσε ενεργητικό ρόλο στο Κοινοβούλιο. Οι υποφαινόμενοι και ε, από πολιτικής απόψεως έχει κάθε ε, ε, δικαίωμα αλλά και κάθε υποχρέωση να φέρει σε πέρας και να διαλευκάνει αυτήν την υπόθεση. Ε, τον, τους προηγούμενους ε, μήνες ξεκινήσαμε ε, ένα διάλογο με την περιφέρεια της Καμπανίας και επίσης τα τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει και διάλογος με την Κομισιόν. Δεν υπάρχει τίποτα περίεργο ή αξιοθαύμαστο στην προκείμενη περίπτωση μετά από σειρά ετών που είτε δεν αναλήφθηκα μία δράση είτε οι δράσεις που αναλήφθηκαν δεν οδήγησαν προς σωστή κατεύθυνση ε, και οδηγηθήκαμε στην γνωστή κατάσταση του 2007 ε, άλλαξαν κάπως ε, τα πράγματα Ήδη ο ε, επαρχιακός υπεύθυνος έχει έρθει τρεις φορές ε, στις ε, Βρυξέλλες και έχει ήδη ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος που είχε αναφέρει σε μια ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών. Το πρόγραμμα στερεών αστικών αποβλήτων έχει υποβληθεί και έχει διορθωθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκριθεί μέχρι τις 30 Απριλίου. Έχει ήδη όμως ε, ξεκινήσει η πίεση του. Ε, έχουν ε, ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες διαγωνισμού για το Σαλέρνο. Επίσης οι ίδιες διαδικασίες για την Νότια Νάπολη. Έχουν ξεκινήσει τέσσερις, τέσσερα κέντρα διαλογής, 30 κλασικές πλατφόρμες και βεβαίως χαίρομαι και μια σειρά σειρά άλλων ε, στοιχείων που χαίρομαι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει δεχτεί ε, όλα τα στοιχεία αυτά. Επίσης έχουν, έχουν υπάρξει συμφωνίες με πέντε επαρχίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη να υλοποιούν προγράμματα εν αναμονή της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος μετά από την συμφωνία, μετά από την έγκριση του συνολικού σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπότιτλοι Authorwave 12 με 24 μήνες σύμφωνα με την κυρία Μπουτσέλα και σύμφωνα με αυτά που είπε ενώπιον ε, τη ε, επιτροπή μα στην Ακρόαση ε, χρειάζονται έτσι ώστε να διαλεγούν όλα τα συσσωρευμένα απόβλητα. Όπως είπε και ο επίτροπο, δεν μας ενδιαφέρει να δοθούν, να επιβληθούν νέα οικονομικά πρόστιμα. Μας ενδιαφέρει επίσης να μην εγχειρηματοποιηθεί η συζήτηση αυτή. Ε, δεν θέλουμε ε, αυτή η συζήτηση να αφορά ε, μονάχα τις πολιτικές αρχές. Εάν θέλουμε πραγματικά η συζήτηση αυτή να αφορά την καμπανία, εάν θέλουμε να, γίνουν, να γίνει ένας πραγματικός διάλογος, τότε μπορούμε να οδηγηθούμε πραγματικά το Φεβρουάριο σε μια κοινή συζήτηση, γιατί διαφορετικά θα χάσουμε χρόνο, θα χάσουμε πολύτιμες προσπάθειες. Πρόεδρος, δεν διέκοψα την ε, κυρία Ματσόνη. Ε, ε, θα, ήθελα όμως να σας παρακαλέσω πρώτον να μην ξεπερνάτε το χρόνο σας και δεύτερον να μην τρέχετε με τον τρόπο αυτό. Να, να μιλάτε με ένα ρυθμό φυσιολογικό έτσι ώστε να επιτρέπετε στους διερμηνείς να, κάνουν, να παρακολουθούν την συζήτηση. Ο κύριο Πυρίλο, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, η βαθιά κρίση η οποία αφορά τη διαχείριση διαχείριση των αποβλήτων ε, στην ε, περιοχή τη ε, Καμπανίας Βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει σημαντικέ επιπτώσει στην ποιότητα ζωή των πολιτών. Ω πολιτικοί έχουμε την υποχρέωση και την ευθύνη να παρέμβουμε έτσι ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και βεβαίω να κρούσουμε και τον κόδωνα του κινδύνου στι τοπικέ αρχέ, έτσι ώστε να εγκρίνουν αξιόπιστα προγράμματα που θα επιτρέψουν στην Καμπανία να εξέλθει από αυτή τη βαθύτατη κρίση. Είναι αλήθεια ότι πολλή λόγος έγινε ε, για το πρόβλημα αυτό και πρέπει κανείς να ξέρει πώς έχουν τα πράγματα. Η Επιτροπή της ε, ε, Καμπανίας ήδη από το 2010 είχε ε, δεσμευτεί να υποβάλει πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιεί το άμεσα και το οποίο όμως παρεπέμφθη τώρα στον Απρίλιο του 2011. Σε λίγο η κατάσταση δεν θα μπορεί πλέον να τη διαχειριστεί κανείς και βεβαίως υπάρχουν, ε, εξακολουθούν να υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κερδίζουν χρήματα ε, από την κρίση η απόφαση να ε, δοθεί πλήρης αρμοδιότητα στις επαρχίες και στις περιφέρειες για την διαχείριση των αποβλήτων είναι μια απόφαση την οποία δεν συμμεριζόμαστε. Ε, μονάχα οι μικρές κοινότητες ε, και οι μικροί δήμοι είναι σε θέση να δώσουν στοχευμένες και αποτελεσματικές λύσεις. Ε, παρά την ε, προσπάθεια δεν έχουμε ικανά αποτελέσματα, ικανοποιητικά αποτελέσματα ε, όσον αφορά την κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είχαμε αποκεντρωμένη διαχείριση από τις κοινότητες και τους Δήμους, τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα. Τώρα βλέπουμε όμως ότι παίρνουμε από τα χέρια των Δήμων κάθε αρμοδιότητα και τη βάζουμε στα χέρια των επαρχιών και των περιφερειών. στο Τερτσίνιο και στην ε, Κάβα Πιτιέλο ε, ζητήσαμε να μην υπάρξουν κέντρα ε, διότι πρόκειται για σημεία προστατευόμενα η, περιμένουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στο πρόγραμμα το οποίο έχει υποβάλει η περιφέρεια της Καμπανίας. Ευχαριστώ πολύ εξ ονόματος των φιλελευθέρων η κυρία Αλφάνο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Παρά την προπαγάνδα της Ιταλικής κυβέρνησης ε, που διαψεύστηκε άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πράγματα δεν έχουν προοδεύσει και δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και υπάρχει ε, μία σταθερά. Δηλαδή ότι εξακολουθούν να ζουν και να πεθαίνουν μέσα στα σκουπίδια οι κάτοικοι της ε, Καμπανίας. Ε, και η δεξιά και η αριστερά έχουν πάρα πολύ σημαντικές ευθύνες και το βέβαιο είναι ότι δεν μπορεί τελικά να αποδοθεί η ευθύνη εις τους πολίτες γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βγούμε από την κατάσταση ή ε, τα σημεία, οι εγκαταστάσεις ε, καύσης ε, που έχουν χρηματοδοτηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Είναι επιβλαβής για την υγεία και βεβαίως δεν μπορούν να υποκατασταθούν από άλλες λύσεις οι οποίες σέβονται τη ζωή των πολιτών, σέβονται το περιβάλλον. Βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε είναι ότι ε, η μαφία ε, που εκμεταλλεύεται τα σκουπίδια δεν αφορά μονάχα τον Νότο, δεν δρά μονάχα στον Νότο, αλλά κυρίως το Βορρά από τα τελευταία χρόνια. Το ζήτημα είναι ότι εξακολουθούν οι πολίτες να είναι όμοιροι, ε, εξακολουθούν να υφίστανται ε, ε, λύσεις οι οποίες τελικά δεν οδηγούν πουθενά. Οι πολίτες εξακολουθούν να ζουν σε στρατοκρατούμενες περιοχές. Τι προτίθεστε να κάνετε έτσι ώστε να βοηθήσετε την περιοχή. Με ποιο τρόπο προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 260 της συνθήκης κατά της Ιταλίας απαιτώντας επιβολή χρηματικών κρατικής ποινή και με ποιο τρόπο προτίθεται να ελέγξει τις κρατικές επιδοτήσεις και τον τρόπο χρήσης τους. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από τις ιστορίες των συναδέλφων του έλτε επανέρχομαι σε πρακτικά θέματα. Είναι γεγονός ότι έγινε προσφυγή και καταδίκη πολύ σωστά της Ιταλίας. Η Ιταλία δεν τήρησε τις προθεσμίες. Προφανώς το σχέδιο το έδωσε η περιφέρεια αλλά μετά δεν πήγε παραπέρα. Έτσι είναι ίδια η κατάσταση. Και βέβαια δημιουργείται η εντύπωση ότι οι υπεύθυνοι συνεχίζουν να τραβάνε τα πράγματα μέχρι να δημιουργηθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά ισχύουν οι νόμοι για την έκτακτη ανάγκη στην Ιταλία, πάνω εκεί πάνω σε αυτή τη βάση λαμβάνονται οι αποφάσεις, όλα τα άλλα ακυρώνονται. Όταν είναι πολλά τα σκουπίδια στο δρόμο μαζί με βιομηχανικά απόβλητα από βορρά και νότο, τότε γρήγορα κάπου πάνε χωρίς καμιά ασφάλεια σε χωματερή, χωρίς ε, καμία πρόληψη, κανένα μέτρο προστασίας. Δεν είναι συζήτηση μεταξύ Ιταλών αγαπητοί μου Ιταλοί συνάδελφοι, αυτή είναι μια συζήτηση όπου δεν τηρείται το ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν εφαρμόζεται. Αν αυτές οι μεθοδεύσεις επεκταθούν και σε άλλες χώρες μέλη, αυτό θα έχει πανευρωπαϊκές επιπτώσεις. Δεν είναι ε, μια ιδιαίτερη περίπτωση, ε, δεν είναι κάτι συνηθισμένο, είναι σκάνδαλο. Δεν είναι δυνατόν να τα στέλνουμε από εδώ και από εκεί και μετά να απειλούμε με την αστυνομία τους διαμαρτυρώμενους πολίτες που δεν θέλουν με τα οικιακά απόβλητα να πετάγονται και τα βιομηχανικά στις χωματερές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να υπάρξουν απτές, αισθητές επιπτώσεις, συνέπειες είναι καλό που δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται όπως παλιά τα μέσα για την ε, αντιμετώπιση του θέματος, διότι πρέπει να νιώσει στο πετσί της η Ιταλία τις συνέπειες, γιατί εδώ πρόκειται για πολύ ε, σημαντικό και ορθολογικό και λειτουργικό ευρωπαϊκό δίκαιο που δεν τηρείται και πρέπει να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο ε, κύριος Χίγγινς δεν είναι εδώ, επομένως θα δώσουμε το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Ρώση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόγραμμα αποκομιδής ε, των, ε, των αποβλήτων βεβαίως θα πρέπει να περιέχει διάφορα στοιχεία υπενθυμίζω ότι ε, ε, η, δικιά σας, ε, ο δικός σας πολιτικός σχηματισμός των Πρασίνων που είχε και προκαιρού ακόμα και υπουργό δεν έκανε τίποτα. Επομένως να μην λέμε ότι θέλουμε. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση είναι τραγική. είναι γεγονός επίσης ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε για δικαιολογίες. τώρα το να λέει κανείς ότι ο Βορρά ευθύνεται για την κατάσταση στο Νότο ε, βεβαίως ε, ε, δεν ισχύει. Γνωρίζομαι ποιες είναι οι παράνομες πρακτικές οι οποίες σχετίζονται με την, με την αποκομίδη των σκουπιδιών. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μέσω των, της ψήφου τους οι κάτοικοι της Καμπανίας όπως έκαναν σε τελευταίες εκλογές να αλλάξουν τους πολιτικούς υπευθύνους. Ευχαριστώ πολύ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η κρίση των αποβλήτων στην περιοχή της Νάπολης τώρα διαρκεί 14 χρόνια. Ε, έχουν γεμίσει οι χωματερές, μπλοκάρονται εντωμεταξύ και από τους πολίτες που δυσπιστούν απέναντι σε οποιοδήποτε σχέδιο. Αυτό εξηγείται, διότι σε πολιτικό επίπεδο δίνονται τώρα πολλές υποσχέσεις που δεν τηρούνται σχεδόν καθόλου. Η διαχείριση του προβλήματος μέχρι τώρα ε, στηρίχθηκε σε μεταβατικές λύσεις προσωρινές. Ε, ε, υπήρξαν ειδικά προγράμματα που δεν μπόρεσαν ούτε καν να ενημερώσουν τις τοπικές κοινότητες και από την άλλη πλευρά ε, αυτές οι καταστάσεις έγιναν καθημερινότητα στην Ιταλία. Πολύ πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δεν δίνεται καμία σημασία στη διαλογή, στην ανακύκλωση. Έτσι λοιπόν δημιουργείται πρόβλημα και στην περιβαλλοντική συνείδηση. Η Καμπανία είναι μια μολυσμένη περιοχή, η καρκίνη έχουν και τα αναπνευστικά νοσήματα στην περιοχή αυτή είναι πολύ πάνω από τον Ιταλικό μέσον όρο. Άρα πρέπει κατεπηγόντως να εξευρεθούν και να εφαρμοστούν λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ οι υπόλοιποι γεγραμμένοι. Θα αρχίσουμε με την κυρία Ριβελίνη για δύο λεπτά. Τον κύριο Ριβελίνη, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, το, ε, τους συναδέλφους που μου ανέθεσαν ε, να μιλήσω, αλλά πρέπει να σας πω ότι ήδη στην καμπανία έχουν ήδη ξεκινήσει εξαιρετικά θετικές διαδικασίες. Σύμφωνα με το τέος 200, άρθρο 260 του κανονισμού, τα οικονομικά πρόστιμα δεν υπάρχει λόγος πλέον να εφαρμόζονται. Έχουμε μια καινούρια ε, περιφερειακή Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει μια νέα πολιτική όσον αφορά ε, την ε, διαλογή των σκουπιδιών καθώς επίσης και πρωτοβουλίες για την μείωση της παραγωγής αποβλήτων. Στο Σαλέρνο έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για αποτεφρωτήρα και στην Δυτική και Νότια Νάπολη έχουν προχωρήσει πολλοί διαγωνισμοί για αντίστοιχες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης μείωση των ε, παραγωμένων ε, αποβλήτων, ε, διαλογή των αποβλήτων, καθώς επίσης και δημιουργία ειδικών χιτά και στους τρεις τομείς τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Βεβαίως και οι τέος αρχές που διοικούσαν την καμπανία, που ήταν αρχές αριστερές και πρασίνων, ευθύνονται για την κατάσταση. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει την ε, Καμπανία. Ε, θα πρέπει να εργαστεί με την Καμπανία και όχι κατά ε, της Καμπανίας. Πρέπει κανείς να ξεπεράσει τις πολιτικές του καταβολές. Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα στην Καμπανία γιατί η κατάσταση είναι ιδιαίτερος επίγουσα. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει ο κύριος Ντεματζίστρης για ένα λεπτό μετά από τα ψεύδη της ε, κυβέρνησης ε, Μπερλουσκόνη που το 2008 είπε ε, στην Ιταλική κοινή γνώμη ότι ξεπεράστηκε το πρόβλημα των σκουπιδιών νομίζω ότι η ορθή απόφαση είναι να μπλοκαριστούν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ιταλία μέχρι ότου να ολοκληρωθούν πραγματικά προγράμματα για την αποκομιδή και διαχείριση των σκουπιδιών και όχι σαν αυτό ε, το, του ε, Καλντόρο. Ε, βεβαίως δεν είναι δυνατόν να βάλει κανείς από ε, που προκαλούν καρκίνο, που προκαλούν το θάνατο ή να δημιουργηθούν χιτά σε προστατευμένες περιοχές στους πρόποδες του Βεζουβίου παραδείγματος χάρη. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση όσον αφορά αυτές τις διασυνδέσεις στα ευρωπαϊκά χρήματα, την τοπική ε, διοίκηση, την περιφερειακή διοίκηση, την καμόρα, την μαφία της ε, περιοχές ε, και επομένως να ληφθούν σημαντικές και σοβαρές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Περόνι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κέντρο, κεντρική οργανωμένη και γραφειοκρατική Ευρώπη δεν μπορεί να κατανοήσει τις ε, αποκεντρωμένες διεργασίες ε, στα πλαίσια των κρατών μελών. Η καταστροφική κατάσταση στην Καμπανία ε, κυρίως αφορά ε, την ε, ε, Καμπανία. Και εγώ σαν κάτοικος της Παδανίας στρέφομαι εναντίον όσων ψήφισαν ανίκανους και εγκληματικούς πολιτικούς, τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους και μάλιστα τους ψήφισαν πολλές φορές. Η Παδανία θέλει να βοηθήσει την Καμπανία αλλά δεν αποδέχεται, απορρίπτει με ευδελιγμία τις ε, ε, κατηγορίες. Ευχαριστώ κύριος Μπαλντασάρη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη επίτροπε κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. βεβαίω, με, την, ε, με τα λόγια μου δεν θέλω να αρνηθώ την σοβαρότατη κατάσταση η οποία ε, αποτελεί την, ε, το αποτέλεσμα μιας καταφανούς κακοδιοίκησης κυρίες Λίχτεμπερ και Σόντεργαρντ η κρίση στην καμπανία δημιουργήθηκε και μεγάλωσε λόγω της πλήρους ανικανότητας ε, των περιφερειακών αρχών καθώς επίσης ε, και ε, της αριστερής κυβέρνησης της Νάπολης που είχε και συμβούλους από το κόμμα των Πρασίνων και που δεν κατάφεραν ποτέ να δημιουργήσουν έναν κύκλο ενάρετο όσον αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών ε, σκοτεινές διεργασίες, ε, ανίερες συμμαχίες, πολιτικές, εγκληματικές κλπ. αφορούν το παρελθόν. Αυτός ο κύκλος έχει τώρα ολοκληρωθεί. Θέλω να διασφαλίσω όλους όσους υπέγραψαν τα ψηφίσματα και όλους τους υπολείπους ότι η κατάσταση έχει αλλάξει, ότι ε, οι νέες αρχές έχουν την πολιτική βούληση να ξεπεράσουν τα προβλήματα να ανταπεξέλθουν ε, από ε, οποιαδήποτε προβλήματα υπήρχαν μέχρι τώρα ε, και βεβαίως σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών να ξεπεράσουν αυτό το σύνδρομο που λέει τα σκουπίδια στη δικιά σου αυλή και όχι στη δικιά μου, μακριά από μένα δεν τα θέλω. Έχουν ληφθεί, υπάρχει η πολιτική βούληση και έχουν ληφθεί και οι σημαντικές αποφάσεις ε, δεν είναι δυνατόν και αποτελεί προσπάθεια χειραγώγης της κοινή γνώμης και εγχειρηματοποίησης του προβλήματος αυτό που προτείνει ο κύριος Ντεματζίστρης δηλαδή ε, να σταματήσει η ροή κοινοτικών πόρων προς την ε, περιφέρεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε την κατάσταση, να γυρίσουμε αυτήν την κακιά σελίδα στην πολιετή χιλιετή ιστορία της Νάπολης. Ευχαριστώ πολύ. Σνέλλαρντ για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Ελπίζω η σημερινή συζήτηση να είναι έναυσμα για μεγάλη αλλαγή στο σύστημα αποκομιδής σκουπιδιών στην Καμπανία. Η απόφαση και το, η προτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να εφαρμοστούν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες θα πρέπει να ισχύσουν και για την αποκομιδή και για τη συλλογή των αποβλήτων, διότι οι βλάβες από τις παράνομες χωματέρε πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ξέρω γιατί μιλάω. 20 χρόνια μετά την επανένωση στη Γερμανία ακόμα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα από τι παράνομε και τις ε, κακές συνθήκες ε, αποκομιδής. Όλα αυτά όμως δεν θα πετύχουν αν δεν πιάσουμε τη ρίζα του προβλήματος, ό,τι και να λέμε. Ε, στις ε, διοικήσεις υπάρχουν μαφιόζικες δομές, πρέπει να καταπολεμηθούν για να έχουμε επιτυχία. Και το λέω ειλικρινά, τέσσερις προϋποθέσεις πρέπει να ισχύσουν. Πρώτον, κατάρτιση σχεδίου για την αποκομιδή, υπάρχει αυτό, αλλά και η Κομισιόν πρέπει να βοηθήσει εκεί, θεωρώ. Επίσης, διάθεση δημοσιονομικών πόρων ούτως ώστε να δημιουργηθούν νέες μονάδες ανακύκλωσης κλπ. Σκληρότερες ποινές για την παράνομη αποκομιδή και νομίζω επίσης απευθυνόμενος στην Κομισιόν ότι η Europol και η Eurojust η εισαγγελία, η αστυνομία θα πρέπει να υποστηριχθούν ε, στην καταπολέμηση της παράνομη, του εγκλήματος τα κονδύλια που διατίθενται πρέπει να μην δοθούν μέχρι να ισχύουν οι προϋποθέσεις. Τότε θα συνενέσω να ε, αποδεσμευτούν τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για 1,5 λεπτό. Η κυρία Κόμη, αγαπητέ επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί πρόεδρε, θα ήθελα να επιβεβαιώσω με σαφή τρόπο ότι η κατάσταση των σκουπιδιών στην Καμπανία έχει βελτιωθεί πολύ σε σχέση με το παρελθόν. Η προβληματική είναι περίπλοκη, παρουσιάζει πολλή πλευρά ε, προβλήματα και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να επιληθεί. Ε, προφορικές ε, ερωτήσεις ε, τις οι οποίες μας απασχολούν αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 260 αλλά δεν πρόκειται με την επιβολή χρηματικής ποινής να κάνουμε κάτι αντικειμενικά θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις διαδικασίες επί παραβάση. αυτό που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η υποκειμενική θέση του κράτους. Δεν είναι δυνατόν να πει κανείς ότι η Ιταλία αρνήθηκε την υποχρέωση για συνεργασία. Αντιθέτως, όπως επιβεβαίωσε και ο κύριος Επίτροπος, οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαρκώς σε επαφή με τις αρχές της κυβέρνησης. Ε, βεβαίως ε, είναι ε, ορθές οι κατηγορίες οι οποίες αφορούν την Ιταλία. Όμως θα πρέπει να βοηθηθεί η περιφέρεια έτσι ώστε να μπορέσει να εκπονήσει ένα ορθό σχέδιο. Σε συνέργεια θα πρέπει και, και, και κοντά στην Ιταλία θα πρέπει να βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι θα πρέπει αυτοί που έκαναν πράγματα ή μάλλον που δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι να μην έχουν μικρή μνήμη, να θυμούνται και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Η κυρία Ματέρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν ε, παίρνω τον λόγο σαν εκπρόσωπος της ε, καμπανίας, αλλά ε, για να συμμεριστώ μαζί σας την Ιταλική απάντηση στην κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιφέρεια της καμπανίας αλλά και γενικό ειδικότερα το Ιταλικό κράτος ε, προβλέπουν την δημιουργία ενός ευρύτερου ε, ε, δικτύου αποκομιδής και ανακύκλωσης σκουπιδιών βάσει των ευρωπαϊκών αρχών. Υπάρχει το πρόγραμμα 2007-2013 ε, για το 2006 μέχρι 2007 ε, η ε, καμπανία χρησιμοποίησε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την, για την αποκομιδή, την δημιουργία κέντρων υγρής και ξηρής συλλογής ε, ε, σκουπιδιών ε, καθώς επίσης και για τη διαλογή των σκουπιδιών. Όσον αφορά το πρόγραμμα 2007-2013 110 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για την δημιουργία νέων δομών διαχείρισης των σκουπιδιών και 50, 50 εκατομμύρια για τη δημιουργία κοινωνικών, συγγνώμη, Ερευνητικών Κέντρων Αποκομιδής των Σκουπιδιών. Το 2006 έχουν, ε, ήδη το 2006 ε, ε, υπήρξε μείωση των σκουπιδιών στην Καμπανία. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια υλοποίησης των προγραμμάτων βάσει των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γεγονός ότι υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες συμμόρφωσης προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μπορούμε ε, σε άλλη περίπτωση να ε, ε, εξηγήσουμε την κατάσταση αυτή. Κάτσου διά η διαδικασία πλέον. Σε κοιτάς Σε να, λάβω, να αλλάξω την ευκαιρία και να στρέψω προσοχή προς άλλα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες φορές οι κεντρικές αρχές, οι περιφερειακές αρχές δεν δίνουν αρκετή προσοχή στο θέμα των αποβλήτων. Σε μια πόλη της Λιθουανίας κάποιοι επιχειρηματίες ήθελαν να φτιάξουν μια εγκατάσταση ποτέφρος, αλλά ε, παραπλανώντας το κοινό, λέγοντας ότι πρόκειται για μια εγκατάσταση διαλογής αποβλήτων και οι αρχές δεν έδωσαν αρκετή προσοχή σε αυτή την παραπληροφόρηση. Θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή, να παρακαλέσω την Επιτροπή να, δώσει, να προσέξει τέτοιου είδους ε, παραβιάσεις. Όταν δηλαδή οι αρχές δεν ακολουθούν τις ε, διατάξεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ε, διαχείριση των αποβλήτων, των απορριμμάτων. Ευχαριστώ κύριος Γιάρ. Ähm, Κυρία Πρόεδρε, ήμουν ε, σε ένα ταξίδι με την ε, ε, Επιτροπή Αναφερών στην Καμπανία και θα ήθελα να σας πω ότι εκεί το έργο είναι εξαιρετικά δυσχερές γιατί θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα του παρελθόντος, του παρόντος αλλά και του μέλλοντος. Η εντύπωσή μου από αυτό το ταξίδι είναι ότι η διαχείριση των απορριμμάτων την ε, εποχή της επίσκεψης λύθηκε εν μέρη με ε, τη βοήθεια του στρατού και τα, τελικά τοποθετήθηκαν τα απορρίμματα παράνομα σε τερέσε. Όσον αφορά τώρα το μέλλον, θεωρώ ότι η πρώτη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σωστή και δίκαιη. Εάν η περιφέρεια υποβάλει ένα λογικό σχέδιο διαχείριση των απορριμμάτων, θα αποδεσμεύσει τα κονδύλια Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις τοπικέ αρχές να πράξουν κάτι τέτοιο και θα ήθελα να επαναλάβω ότι από τη δική μου οπτική γωνία, η Επιτροπή και εμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δεν ενδιαφερόμαστε την επιβολή ε, προστήμων, αλλά θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων στην περιφέρεια της ε, Καμπανίας. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Ριβελίνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ενδεχόμενο εμπλοκή των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι αυτοί που αφορούν την βελτίωση του υπεδάφους. Πώς είναι δυνατόν να ε, σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να μπλοκαριστούν αυτοί οι πόροι. Ζητώ από τους ε, πολιτικούς, κυρίως αυτούς που εκλέγονται στην περιοχή της Καμπανίας, να μην παρασυρθούν από την πολιτική τους φρενίτιδα και να μην είναι κακοί για την ίδια τους την, ε, ε, την περιφέρεια ε, και να μην θεωρούν ότι μπορούν να πούν οτιδήποτε αρκεί να προωθήσουν τον εαυτό τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις που εκφράσατε. Τρία-τέσσερα θέματα θα με απασχολήσουν. Πρώτον, αυτό που επανειλημμένα πολύ θέσατε. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Δεν λύνεται γρήγορα. Υπήρξαν κάποιες θετικές εξελίξεις, αλλά προφανώς ακόμα χρειάζεται συστημική απάντηση στο υφιστάμενο πρόβλημα δεν είναι εύκολο, αλλά απαραίτητο όσο δεν πάει άλλο. Υπ' αυτή την έννοια, ο εταίρος μας για στην εξέβρεση λύση είναι η Ιταλία βέβαια, αλλά η συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές αναμφίβολα χρειάζεται εδώ. Οπότε προσβλέπω ειλικρινά στην αξιολόγηση του νέου σχεδίου διαχείρισης σχέδιο προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων. Ελπίζομαι να είναι αυτό που θέλουμε. Θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες μου και σας διαβεβαιώνω ότι η αξιολόγηση θα γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να αντιμετωπιστεί με ισότιμο τρόπο η Ιταλία όπως και άλλες χώρες μέλη γιατί είναι σημαντικό να διατηρείται εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών. Όταν μιλάμε λοιπόν για το χειρισμό αυτού του ζητήματος, η προσέγγιση μου θα μπορούσε να διατυπωθεί με τέσσερις λέξεις. Θέλω να είμαι ε, να, να επικουρήσω με αυστηρό τρόπο και να είμαι αυστηρός επικουρώντας. Η ιδέα λοιπόν όπως είπατε και αρκετοί από εσάς είναι η επίλυση των προβλημάτων. Αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος όμως τα προβλήματα θα πρέπει να επιληθούν μέσα από την επιβολή προστήμων. Είναι καθήκον μου να τα επιβάλλω, δεν γίνεται αλλιώ. Κάνω ό,τι είναι δυνατόν ειλικρινά σε συνεργασία με τις Ιταλικές αρχές ώστε να εξευρεθεί η κατάλληλη λύση και ελπίζω ειλικρινά ότι θα τα καταφέρουμε γιατί σε τελευταία ανάλυση μιλάμε για την υγεία των Ιταλών και του περιβάλλοντος τους. Το επόμενο θέμα αφορά την ε, οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα που πρόσφατα εγκρίθηκε και αυτή η οδηγία είναι ξεκάθαρη. Προβλέπει ότι κάθε κράτος θα πρέπει να ε, εισαγάγει η ιεράρχηση των αποβλήτων. Ο το καλύτερο απόβλητο δεν είναι απόβλητο. Θα πρέπει λοιπόν να ε, υπάρξει ε, νέα παραγωγής ενέργειας, ανακύκλωση, παραγωγή ενέργειας και ε, χωματερή ηχητά, αν δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή ε, είναι μια εικόνα που αφορά την αποτελεσματικότητα των κρατών μελών, είναι από την έκθεση που έχουμε. Αφορά τις τάσεις του ΧΙΤΑ στα αστικά απόβλητα, γιατί από τα αστικά απόβλητα έχουμε τα καλύτερα στοιχεία πέντε κράτη-μέλη, πιστέψτε το, σε πέντε κράτη-μέλη η χιτά είναι κάτω από το 5%, κάτω από το 5% των ε, αστικών αποβλήτων. Αλλά 7 κράτη-μέλη ε, σε 7 κράτη-μέλη οι χιτά, οι χωματερές είναι πάνω από το 80% των αστικών αποβλήτων. Οπότε βλέπετε μεγάλες διακυμάνσεις στην κατάσταση στην Ευρώπη στο χειρισμό αυτών των θεμάτων. Και προφανώς αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Θέλουμε. Αλλά αν δείχνει κάτι η εικόνα αυτή, γιατί είναι μια εικόνα από το 1995 μέχρι το 2007, αν θέλουν οι χώρες να αλλάξουν, θα αλλάξουν. Αν οργανωθούν με το σωστό τρόπο, μπορούν πραγματικά να αλλάξουν. Η Ευρώπη σήμερα μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη έτσι αδερά. Το ένα θεωρεί τα απόβλητα ως πρόβλημα και ένα άλλο μέρος που θεωρεί τα απόβλητα ως μείζωνα ευκαιρία άντλησης πόρων. Και για ε, οικονομικά ωφέλη. Γιατί είναι αλήθεια αυτό. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες που δείχνουν ότι η ανάγκη θα πρέπει να υπάρξουν ε, κρατικές συμβάσεις, δημόσιες συμβάσεις για το ποιος θα αναλάβει τα απόβλητα. Γιατί πολλοί θέλουν να τα αναλάβουν. Η θεμελιώδης ανάγκη είναι να επιλέγονται αυτή εξ αρχή. Δεν γίνεται διαλογή δηλαδή των αποβλήτων από την αρχή. Αυτή είναι η θεμελιώδη πρώτη στη ανάγκη. Τέλο, κάτι τελευταίο που θέλω να αναφέρω αφορά τον συνάδελφο που, το αξιότιμο μέλος που είπε ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με τα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων και αλλού. Στις ε, περιπτώσεις κίνησης διαδικασίας επί παραβάση, τα απόβλητα είναι στο 19% των ε, διαδικασιών. 16, καμιά φορά και λιγότερο. Οπότε βλέπουμε με οριζόντιο τρόπο όλα τα προβλήματα υλοποίησης. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό και θα συνεχίσουμε, σε διαβεβαιώνω και στο μέλλον. Και για να κλείσω, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το καλύτερο. Και εσείς από το Κοινοβούλιο και εγώ ως Επίτροπος Περιβάλλοντος να περάσουμε σε όλη την Ευρώπη το μήνυμα ότι τα απόβλητα συνιστούν ευκαιρία για το μέλλον. Χρειάζεται κατεπηγόντως να αποσταλεί το μήνυμα αυτό δεδομένων των περιορισμένων πόρων που βλέπουμε να έχουμε κάθε μέρα. Αποτελεσματικότητα λοιπόν στα απόβλητα και στους πόρους. Αυτό είναι ο πυρήνας της μελλοντική αποτελεσματικότητάς μας στην Ευρώπη. Αν δεν το πιστεύετε, ελάτε να το συζητήσουμε μετά από 10 χρόνια και σας διαβεβαιώνω ότι έτσι θα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρο στην συνεδρία της Ολομέλειας.